Αγαπητοί συνάδελφοι, να αρχίσουμε. Με το σημείο 14, της ψηφοφορίας. Πρέπει να ζητήσω συγγνώμη για την μικρή αργοπορία, διότι μόλις ε, ήμουν σε μια κοινή δήλωση ανάμεσα στην Επιτροπή και το Συμβούλιο για τον κανονισμό για τα ορυκτά περιοχές ε, συγκρούσεων. Έγιναν πολλά. Καταφέραμε να υπάρχει υποχρεωτική, υποχρέωση μάλλον για τις ε, επιχειρήσεις και ε, upstream και downstream. Καθώς και Κάποιες ε, υποχρεώσεις σχετικά με τις ε, βιομηχανικές πρακτικές. Είναι λοιπόν μια καλή μέρα πιστεύω, ένας κανονισμός ο οποίος είναι προς το συμφέρον των πολιτών, ιδιαίτερα εκείνων που μένουν σε αυτές τις περιοχές. Ε, γι' αυτό λοιπόν αργήσαμε, αρχίζουμε όμως. Όπως γνωρίζετε η πρώτη ψηφοφορία θα είναι δοκιμαστική, έτσι ώστε όλοι να έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τις κάρτες ψηφοφορίας. Άρχεται η ψηφοφορία. Παρακαλώ, να έχω κάποιο πρόβλημα. Μόλις είδα ότι ξέχασα την κάρτα μου στο Στρασβούργο. Όταν θα κάνετε ψηφοφορίε, παρακαλώ, ε, επιτρέψτε μου να ψηφίσω διανατάσεως. Μάλιστα. Ένα μέλο λοιπόν δεν έχει την κάρτα μαζί του, οπότε πρέπει να καταγράψουμε την ψηφοφορία χωρίς κάρτα. Όλα τα υπόλοιπα είναι εντάξει. Δεν υπάρχει κανένα μέλος παραπάνω από κάποια ομάδα. Αρχίζουμε λοιπόν. με την ψηφοφορία για το πακέτο στρατηγικής για το εμπόριο και τις επενδύσεις. Τρία μέρη και τις αιτιολογικές σκέψεις, δηλαδή τέσσερα μέρη. Πρώτο μέρος. Τροπολογία 61. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρο... Συμβαστική τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 68. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 75. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμπληρωματική στην συμβιβαστική 3 έχουμε την 78. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 81 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 83. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 92. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά την 92. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Η δική σας ψήφος. Εκτός μικροφώνου. Η βοηθός μου μόλις μου έδωσε την κάρτα μου. Είναι πολύ αποτελεσματική. Ευχαριστώ. Απορρίπτεται λοιπόν. Τροπολογία 93. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 91. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Την τροπολογία 91. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 94. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 109. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Οι σοσιαλδημοκράτες τι κάνουν. Ξαναρωτώ. Τροπολογία 109. υπέρ. Κατά. Αποχέ. Ενδιαφέρον αυτό ο συνασπισμό. Νομίζω πω εγκρίθηκε, αλλά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 109. Άρχεται. Πέρα. Εγκρίνεται. Αυτό σα είπα κι εγώ. Συμβιβαστική τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 116. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 117. Σε τρία τμήματα. Πρώτο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τρίτο, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 118, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 119, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 120, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 121, υπέρ, Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμπληρωματική είναι η 124. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 122. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 130 υπέρ κατά αποχές Νομίζω πως απορρίπτεται, το ελέγχουμε όμως. 130, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Αμάλιστα. Ένας περισσότερος από το ΕΛΚ. Απορρίπτεται. 131. Υπέρ. Τάβιντ. Θα ήθελα να ζητήσω ψηφοφορία κατά τμήματα. Το πρώτο τμήμα μέχρι το Modern Slavery, δεύτερο τμήμα, and in the meantime. Για την τροπολογία 131, αν όμως δεν έχουν ενημερωθεί οι ομάδες, ε, ας ψηφίσουμε κανονικά. Προφορική λοιπόν τροπολογία, έτσι θα το ερμηνεύσω. Είναι κάποιος αντίθετος με το να κάνουμε χωριστή ψηφοφορία. Ωραία, κανείς, ας το κάνουμε λοιπόν. Τροπολογία 131 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο, υπέρ, Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 138. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 139. Υπέρ. Όχι, με συγχωρείτε, λέει ο Πρόεδρος. Καταπίπτει. Περνάμε στην 142. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. 142. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 148 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 112 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 149 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 151 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 32α. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 153. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Περνάμε στην 238. Υπέρ. Κατά. Ξανά. 238. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω πως εγκρίθηκε, αλλά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 238. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Σχεδόν Εγκρίθηκε λοιπόν 156 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 161 ως ε, συμπληρωματική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 165 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 172 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε 172 πρώτο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία Πέρασε. Εγκρίνεται. 172 δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 173. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 174. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 175. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 177 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 179 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. 180 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 181 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 182 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 183 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 184 υπέρ κατά αποχές Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 184. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 185. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 189 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 188. Όχι, με συγχωρείτε. Τροπολογία 187 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 190 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στο δεύτερο πακέτο. Συμβιβαστική 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οπότε 202 και 203 ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 204 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 205 την ξέχασα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Οπότε 208 που μπορεί να θεωρηθεί συμπλήρωση της συμβαστικής 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Οπότε Συμβαστική 16. Α. Α. Μ. Το δεύτερο τμήμα δεν καταπίπτει. Αναφέρομαι στην 213. Το δεύτερο τμήμα της 213 ψηφίζουμε ως συμπλήρωση στη συμβαστική 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 224 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.33 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίθηκε αλλά για να το δούμε παρακαλώ ψηφίζουμε 2.33 Μακλάκεν ε, παρακαλώ ηλεκτρονικά άρχεται Ορισμένοι δεν θα ψηφίσουν. Πέρας. Μ, εγκρίνεται. 2.36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Καλά, ας ελέγξουμε. Γιατί δεν σηκώνετε όλοι τα χέρια. 2.36 ελέγχουμε. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Όντως. Συμβαστική 43 επέρ κατά αποχές εγκλίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. σημαστική 20 υπέρ κατά Συνήθως η γερμανική ομάδα δεν είναι τόσο γρήγορη, λέει ο πρόεδρος. Ωραία. Συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 267 που μπορεί να εγκριθεί ως ε, συμπλήρωση. Ποιοι υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εδώ έχουμε μία προφορική τροπολογία του ΕΛΚ. Παρακαλώ. Ο Ντάνιελ. Όπως βλέπετε, θέλουμε να προσθέσουμε τη λέξη SWIFT, γρήγορα. Ωραία, να προσθεθεί, προσθεθεί αυτή η λέξη. Έχει κανείς αντίρρηση? Όχι. Ωραία, να την ψηφίσουμε. Α, υπάρχει, υπάρχει μία αντίρρηση. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε τέσσερις. Τέσσερα άτομα. Λοιπόν, κοιτάξτε, συνεχίζω ο Πρόεδρο. Όχι, δεν υπάρχουν αρκετοί. Να ψηφίσουμε. Παρακαλώ, ποιοι είναι υπέρ αυτή τη προφορική τροπολόγηση. Κατά. Εγκρίνεται. Αποχέ, συγγνώμη. Εγκρίνεται. Ωραία. Δύο ογδόντα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.83 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.82 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.91 υπέρ. Κατά αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά παρόλα αυτά έλεγχος για την 2.91 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 26 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρακόσια Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 307 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 308 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 309 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 310 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3.11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται νομίζω αλλά έλεγχος ε, ελέγχουμε την 3.11 άρχεται πέρας εγκρίνεται συμβαστική 28 υπέρ Υπέρ λοιπόν της συμβαστικής 28 κατά αποχές εγκρίνεται. 3.17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3.32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3.33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3.35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ως συμπλήρωση για την 22 θα μπορούσε να είναι η 373 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 23. Α, θέλετε να ελέγξουμε. Καλώς. Ελέγχουμε την 373 ως συμπλήρωση στη συμβαστική 22 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Ωραία. Λοιπόν, συμβαστική 23 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 24 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 3.53 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 40 υπέρ, κατά αποχές δεν κρίνεται. 3.54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. 3.54 άρχεται. Πέρας. Μα Σα παρακαλώ, να σηκώνετε τα χέρια σα. 33 συμβαστική υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Οπότε περνάμε στην 364. Και η DV18 είναι ταυτόσιμη. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 365 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 366 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 367 και 368 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 369 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 370 υπέρ κατά αποχές. Για να ελέγξουμε την 370 παρακαλώ άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 371 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 372 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι και αυτή απορρίφθηκε, αλλά για να δούμε. Ελέγχουμε την 372. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 379 υπέρ κατά αποχές μάλλον απορρίπτεται αλλά για να δούμε άρχεται πέρας απορρίπτεται Συμβαστική 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 387 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 388 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 389 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 391 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 392 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 393 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 395 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 394 υπέρ κατά αποχές για να ελέγξουμε την 394 άρχεται πέρας απορρίπτεται 396 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 397 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 399 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 400 άρα ελέγξουμε καλά ελέγχουμε την 399 άρχεται Πέρας. Εγκρίνεται. 400. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 402 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 38 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 39 υπέρ. Κατά αποχές. Ενδεχόμενη Δεχόμενη συμπλήρωση. 4-12 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 4-14 υπέρ κατά άποχες για να ελέγξουμε την 4-14 άρχεται πέρας εγκρίνεται να περάσουμε στο τρίτο τμήμα Αρχίζει με την συμβιβαστική α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Τροπολογία 18. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 23. Παρακαλώ, έλεγχο θέλετε. Ελέγχουμε την 22. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 23. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τραπολογία 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 40 υπέρ κατά αποχές νομίζω εγκρίνεται αλλά σε ελέγξουμε. Τροπολογία 40 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Τι γίνεται με τους σοσιαλδημοκράτες, μάτια να ψηφίζουν. Εγκρίνεται μάλλον, αλλά ας το κάνουμε σωστά. 41. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 42. Υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 43. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική F υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 47. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική G. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται.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 Εγκρίνεται. Η 1 και η 2. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 4. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω απορρίπτεται. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 7. Άρχεται.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 εγκρίνεται. Άφετ 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην γνωμοδότηση ΔΕΒΕ. ΔΕΒΕ 5 ως ε, συμπλήρωση στην συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ελέγχουμε. Ελέγχουμε την ΔΕΒΕ 5. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύε 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύε 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύε 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύε 14. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην έμπλη έμπλη 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. έμπλη 18 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε ηλεκτρονικά την έμπλη 18. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Ήτρε τώρα. Ήτρε 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την Ήτρε 20. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Ήτρε 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ήτρε 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ήτρε 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω απορρίπτεται. Ας ελέγξουμε όμως. Ήτρε 21. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Ήτρε 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ήμκο. Ήμκο 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ήμκο 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω εγκρίνεται. Ελέγχουμε. Ήμκο 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ινικό 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Οι σοσιαλδημοκράτες τι κάνετε με την 4. Εγκρίνεται. Ινικό 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ινικό 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές Νομίζω εγκρίνεται. Ελέγχουμε την ΙΜΚΟ 13. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. ΙΜΚΟ 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. ΙΜΚΟ 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Κανείς δεν ασχολείται. Ήμκο 22. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην Επιτροπή Γεωργίας. Άγκρι. Άγκρι 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άγκρι 8 υπέρ, κατά, άποχες. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ να βλέπω χέρια. Άγκρι 8, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται. Μεγάλη πλειοψηφία. Άγκρι 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 20 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 28 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 33 υπέρ. Κατά. Αποχές Νομίζω απορρίπτεται. Ας ελέγξουμε. Άγκρι 33. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Άγκρι 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άγκρι 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άγκρι 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Άγκρι 42. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Άγκρι 43. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω εγκρίνεται. Ας ελέγξουμε για να είμαστε σίγουροι. Άγκρι 43. Πέρας. Απορρίπτεται. Και με αυτό περνάμε στην τελική ψηφοφορία αυτής της πολύ ωραίας έκθεσης. Φυσικά η ηλεκτρονική ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 30 ψήφοι υπέρ. Συγχαρητήρια κυρία Μπεγκίν. Ε, ε, Μάλιστα. Και επειδή μας αρέσει τόσο πολύ να ψηφίζουμε, έχουμε κι άλλα. Και συνεχίζουμε αμέσως με αυτά. Με την ψηφοφορία της έκθεσης της κυρίας Φορέντσα για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, ανθρώπινα δικαιώματα και την εταιρική ευθύνη. Συμβιβαστική τροπολογία 3. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. απόχέ, Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Κατά. απόχέ. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 63. Υπέρ. Κατά. αποχέ, Εγκρίνεται. Τροπολογία Ντέβε για την παράγραφο 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 175 και 176. Ταυτόσιμες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. 175 και 176. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ε, 153. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 154 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω εγκρίνεται. Ας ελέγξουμε. 154. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 12, ε, παράγραφος 12 των γυναικών υπέρ κατά, κατά Mm. Ορίστε. Ναι. Το δεύτερο τμήμα της 155. Πρέπει να το ψηφίσουμε και αυτό. Ποιος είναι υπέρ του δεύτερου τμήματος της 155. Κατά αποχές απορρίπτεται. Λοιπόν, Επιτροπή Γυναικών παράγραφος 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Επιτροπή Γυναικών 14 4 ε, συγγνώμη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογία 51 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 90 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε άρχεται η ψηφοφορία επί της 90 και πέρας και εγκρίνεται συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 2 υπέρ πως είπατε εντάξει εντάξει λοιπόν έλεγχος 81 άρχεται Πέρας. Ε, νομίζω απορρίπτεται. Mm. Εντάξει. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 16. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 164 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 136 το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Καλώς, ελέγχουμε το δεύτερο τμήμα της 136. Άρχεται. Πέρας. Απόλυτα. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται, απορρίπτεται. Συμβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 3 της Επιτροπής Γυναικών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ναι, ναι, βεβαίως να ελέγξουμε. Παράγραφος 3 ε, της Επιτροπής Γυναικών ε, έλεγχος άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται, εγκρίνεται. Συμβαστική 9. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στο δεύτερο τμήμα τώρα. Συμβαστική 13. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 201 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 185 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 186 δύο τμήματα. Το πρώτο παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 187 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 188 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 191 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 200 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 159 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 192 υπέρ κατά αποχές έλεγχος της 192. Άρχεται. Ε, κάποιος, α, εν πάση λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Επιτροπή Γυναικών, παράγραφος 15, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται Επιτροπή Γυναικών 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται να ελέγξουμε ΦΑΜ 17 ελέγχουμε άρχεται πέρας απορρίπτεται ΔΕΒΕ παράγραφος 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έμπλ παράγραφος 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έμπλ παράγραφος 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έμπλ παράγραφος 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οπότε καταπληκτούν 2 και περνάμε στην 162. Υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπλ παράγραφος 26. Υπέρ. Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Συγγνώμη, συγγνώμη. ΔΕΒΕ ε, παράγραφος 7, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δύο ταυτόσημες. Η 111 και η έμπλη παράγραφος 28, υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Έμπλη παράγραφος 29, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται και τροπολογία 2 αναελέξουμε ωραία ελέγχουμε την έμπλ παράγραφος 29 άρχεται πέρας απορρίπτεται 2.19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Περνάμε στο τρίτο τμήμα. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12 ε, υπέρ κατά α με συγχωρείτε με συγχωρείτε τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έλεγχος καλά ελέγχουμε την 20 άρχεται πέρας εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 δύο τμήματα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστή α μάλιστα ελέγχουμε την 29 άρχεται πέρας απορρίπτεται όπως είχα πει. Συμβαστική C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Φα με τη λογική σκέψη ε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Με τη λογική σκέψη H γυναικών υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 32 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Οπότε το F πέφτει. 33 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 46 <clears throat> υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αιτιολογική σκέψη α άφετ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αιτιολογική β άφετ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ετολογικη σι από την άφετ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται για την ιδεολογική ιδέα από την ΑΦΕΤ ε, έχει ζητηθεί κατά τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα, ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Αιτιολογική ε άφετ υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Αιτιολογική εφ άφετ υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Παράγραφος 1 άφετ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 2 άφετ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται καλά να ελέγξουμε την 4 Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. πέντε υπέρ. Κατά. Αποχές. Οι φιλελεύθεροι τι ψήφισαν. Λοιπόν, επαναλαμβάνω τους βοήθεια. την πέντε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άφετ Ετολογική αναφορά 1 υπέρ κατά ε, ε, εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα τελική ηλεκτρονική ονομαστική ψηφοφορία άρχεται και πέρασε και συγχαίρουμε. 30 ψήφοι υπέρ. Συγχαρητήρια. So, Helmut. Helmut, έχεις κάτι διαδικαστικό να πεις. Αγαπητοί συνάδελφοι, ησυχία. Μία πρόταση για την Επιτροπή έχω. Ακριβώς επειδή η Ολομέλεια του Ιουλίου ε, θα εξετάσει την έκθεση που ψηφίσαμε σήμερα, δεν είναι στην ημερήσια διάταξη. Προτείνω λοιπόν εμεί ως Επιτροπή να προτείνουμε να γίνει ανταλλαγή απόψεων, διότι και οι δύο εκθέσεις είναι σημαντικές. Θεωρώ λοιπόν σημαντικό να ζητήσουμε στην διάσκεψη Πρόεδρων Επιτροπών να συμπεριληφθεί ε, και, στην... και να συμπεριληφθεί η συζήτηση και για τις δύο εκθέσεις. Μάλιστα. Πρέπει να το ζητήσετε και ως πολιτική ομάδα, αλλά συμφωνώ με αυτό που λέτε. Ωραία. Η εισηγήτρια θέλει να προσθέσει κάτι. Ναι, κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ με την πρόταση που μόλις τώρα έκανε ο Χέλμουτ Προβλέπονται δύο σύντομες μόνο παρουσιάσεις για τις δύο αυτές εκθέσεις. Συνεπώς θεωρώ και εγώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε πλήρη συζήτηση και για τις δύο εκθέσεις. Ή έστω μια κοινή συζήτηση που να καλύπτει και τις δύο εκθέσεις. Ευχαριστώ. Yeah, I support the position of my colleague. Ναι, συμφωνώ και εγώ με τη συνάδελφο. So, ich würde vorschlagen... Λοιπόν, προτείνω επειδή έχουμε καθυστερήσει να ε, τη συζήτηση για την ε, παρακολούθηση δραστηριοτήτων ομάδων, επειδή δεν είναι και τόσο ενδιαφέρουσα, να την αναβάλουμε για τον Ιούλιο. Υπάρχουν αντιρρήσει. Όχι. Να αναβληθεί το θέμα για την παρακολούθηση δραστηριοτήτων ομάδων για την επόμενη συνεδρίαση, διότι έχουμε καθυστερήσει. Συμφωνείτε. Περνάμε στο σημείο 17. Είναι ένα περισσότερο τεχνικό ζήτημα προσαρμογής των παραχωρήσεων στα πλαίσια της προσχώρησης της Κροατίας μια ανταλλαγή επιστολών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουρουγουάης. Θα δώσω αμέσως το λόγο στον εισηγητή Πάμπλο Ζάλπα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είναι η πρώτη έκθεση που συζητάει η Επιτροπή μας ε, Διεθνούς Εμπορίου για προσαρμογή συμφωνιών με τρίτες χώρες λόγω της προσχώρησης στην Ένωση της Κροατίας. Η προσχώρηση αυτή ε, επεκτείνει και την Τελωνιακή Ένωση. Οι, νόρμες, οι προδιαγραφές ε, του ΠΟΕ είναι ε, Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει διαπραγματεύσεις με τα μέλη του ΠΟΕ που έχουν δικαιώμα διαπραγμάτευσης σε σχέση με το κοινό δεσμολόγιο μετά την προσχώρηση της Κροατίας. Προφανώς πρέπει να υπάρξει αυτή η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ανατολική Δημοκρατία της Ουρουάης. Είναι αναγκαίο λοιπόν να δούμε κάποια αντισταθμιστική προσαρμογή του ε, ε, ισχύοντος δασμολογίου. Οπότε θα προσαρμόσουμε για το κοινό δασμολόγιο των 28 αυτά που υπήρχαν στο κοινό δασμολόγιο των 27 με ε, κάποιες ε, προσαρμογές ε, συγκεκριμένα με κάποια αύξηση των ποσοτήτων βοήου κρέατος. Αυτό είναι αναγκαίο για να επικυρωθεί η συμφωνία. Και ως εισηγητής της Επιτροπής μας, συγγνώμη, ως εισηγητής της Επιτροπής για τη σχέση με το Μέρκοσουρ, Πιστεύω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε με την απόφαση του Συμβουλίου. Όπως ε, και το Συμβούλιο και η Επιτροπή πρέπει και εμείς να δράσουμε για να γίνει αυτή η αναθεώρηση των δασμολογικών παραχωρήσεων. Αυτό αποδεικνύει το κλίμα άλλο που έχουμε με τον ε, εταίρο μας στην Ουρουάη και πόσο σημαντικό είναι να παραχωρήσουμε στα κράτη-μέλη του Μέρκοσουρ αυτά που τους αρμόζουν. Αυτό το είχαμε και τον ε, προηγούμενο μήνα όταν συμφωνήσαμε σε μια συμφωνία εταιρικής σχέσης με το Μερκοσούρ. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές για να προχωρήσουμε και τις γενικότερες εμπορικές διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Δεν νομίζω να θέλει κανείς να πάρει το λόγο, έτσι δεν είναι. Εξ ονόματος Νίκολα Ντάντε να πω ότι υποστηρίζουμε την θέση του εισηγητή. Πρόκειται για ένα τεχνικό ζήτημα και νομίζω ότι θα πρέπει να εγκριθεί το συντομότερο δυνατό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Πολύ σύντομα και εγώ να πω ότι συμφωνώ. Είναι μια τεχνική απλώς προσαρμογή αυτή που συζητάμε αυτή τη στιγμή και προφανώς συμφωνούμε πλήρως με τον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει κάποιο σχόλιο. Όχι. Ο εισηγητή όχι, τίποτα. Σας ευχαριστώ απλώ. Πολύ ωραία. Η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών 22 Ιουνίου στι 6 και ας δούμε αν θα ψηφίσουμε μετά τον Ιούλιο ενδεχομένως τον Σεπτέμβριο. Μάλιστα, λοιπόν. Μπορούμε να περάσουμε τώρα στο σημείο 18 της ημερήσιας διάταξης, παρουσίαση μελέτης σχετικά με τον εξυγχρονισμό του εμπορικού πυλώνα της Συνολικής Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεξικού. Γνωρίζετε πώς έχουν ε, οι εξελίξεις με το εμπόριο, με την TTIP αλλά και την TPP, τη Συμφωνία για τον Ειρηνικό. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν στα πλαίσια αυτών των συμφωνιών και η συνολική συμφωνία που έχουμε με το Μεξικό και γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό να συζητήσουμε τον εξυγχρονισμό, τη μεταρρύθμιση της παλιάς μας αυτής συμφωνίας και θα χαρώ πάρα πολύ να ακούσω τα πορίσματα της μελέτης αυτής και έχουμε και δύο καλεσμένους, έχουμε και καλεσμένους, με συγχωρείτε, από το Μεξικό, έτσι δεν είναι. Θα ήθελα λοιπόν να σας καλωσορίσω και τον πρεσβευτή του Μεξικό στην ε, συνεδρίασή μας. Σας ε, ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Δίνω ευθύς το λόγο στον συντάκτη της ε, μελέτης αυτής, τον κύριο Τόρεντ, από το Πανεπιστήμιο της Βαρκελόνης. Έχετε λοιπόν το λόγο. Παρακαλώ. Thank Εκτός μικροφώνου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να διαπραγματευτεί τον εξυγχρονισμό της συμφωνίας αυτής που συνάφθη το 1997. Όταν διαπραγματευτήκαμε και υπογράψαμε τη συμφωνία αυτή το 1997, ήμουνα διευθυντή εξωτερικών εμπορικών ε, σχέσεων στην νομική υπηρεσία του Συμβουλίου. Και με την ιδιότητά μου αυτή ήμουν ένας από τους ανθρώπους που σχεδίασε τη συμφωνία αυτή που καλούμεθα τώρα να εξυγχρονίσουμε. Και χρειάστηκε να εξηγήσω τότε στο Συμβούλιο και στα κράτη-μέλη πώς είχαν τα πράγματα, αλλά και στον πρεσβευτή τότε του Μεξικού, ο οποίος ε, ήθελε να δώσει κάποιες ε, σαφείς ε, απαντήσεις στην κυβέρνησή του όσον αφορά το πολύπλοκο αυτό θεσμικό πλαίσιο το οποίο είχε συμφωνία και ήθελε να λάβει κάποιες απαντήσεις σε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Όταν εμείς συντάξαμε τη μελέτη αυτή και όταν προτίμαζα την παρουσίαση αυτή, ουσιαστικά υιοθέτησα τη στάση που είχα και τότε. Δεν πρόκειται για μια ακαδημαϊκή θεωρητική άσκηση που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ούτε αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να πούμε πράγματα τα οποία θα ήταν ε, ευχάριστα, αν θέλετε, για τους πελάτες μας, αλλά νομίζω ότι μπορούμε πραγματικά να συμβάλλουμε στη χάραξη μιας σωστής εμπορικής πολιτικής, προσπαθώντας να δούμε πραγματικά ποια είναι τα βασικά ζητήματα πολιτικής, τα οποία πρέπει εσείς να αντιμετωπίσετε κατά τη διάρκεια της επραγμάτευσης της συμφωνίας αυτής και για τα οποία θα πρέπει να δώσετε συγκεκριμένη ανάλυση και συγκεκριμένες απαντήσεις. Και πρέπει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμβάλλει ως θεσμικό όργανο που ανέκαθεν ήθελε να επιλύει τα προβλήματα και όχι απλώς να τα κρύβει και να μην στρουθοκαμιλίζει να μην εθελοτυφλεί δηλαδή μπροστά στα προβλήματα αυτά. Θα σας προβάλλω λοιπόν κάποιες διαφάνειες που αναφέρονται στα βασικά ζητήματα πολιτικής, τα οποία θα πρέπει εσείς να λάβετε υπόψη σας. Όταν κάναμε συνεντεύξεις για την ανάλυση της συμφωνίας αυτής, υπήρχαν αυτοί οι οποίοι δεν ήταν κατά, αυτοί που ήταν μάλλον υπέρ και αυτοί που ήταν σαφώς υπέρ μιας φιλόδοξης συμφωνίας. Για την τρίτη αυτή κατηγορία συμμετεχόντων τους ρωτήσαμε αν πραγματικά προτίθανταν να αλλάξουν οτιδήποτε προκειμένου να αλλάξει το θεσμικό καθεστώς αυτό το οποίο επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Μεξικό και μας είπαν δεν θέλουν να αλλάξουν τίποτα. Ουσιαστικά τίθεται το ακόλουθο ερώτημα λοιπόν. Πώς γίνεται μια φιλόδοξη συμφωνία να είναι πραγματικά φιλόδοξη αν δεν αλλάξουμε τίποτα. Προφανώς μ' αρέσει ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, μ' αρέσει πάρα πολύ και ο Γατόπαρδος, το βιβλίο του Λαπεντούζα, καθώς επίσης και η ταινία που έκανε ο Βισκόντι. Δεν νομίζω όμως ότι αυτό το οποίο είπε ο Γατόπαρδος, δηλαδή ότι πρέπει όλα να αλλάξουν προκειμένου να παραμείνουν τα ίδια, αποτελεί εδώ πέρα σωστό γνώμονα όσον αφορά την εμπορική πολιτική. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε εδώ και τα μέλη της Επιτροπής αυτής, αν πραγματικά θέλετε να τροποποιήσετε οτιδήποτε στη συμφωνία αυτή. Πρέπει πραγματικά να δώσετε μια απάντηση στο ερώτημα αυτό, διότι αν δεν αλλάξει τίποτα τότε στη συμφωνία αυτή, τότε και οι επιπτώσεις της συμφωνίας αυτής θα είναι μηδενικές από οικονομικής και πολιτικής πλευράς. Προφανώς υπάρχουν λόγοι που επιβάλλουν τον εξυγχρονισμό της συμφωνίας αυτής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αλλάξει, ο κόσμος έχει αλλάξει, το Μεξικό έχει αλλάξει. Αλλά η διαδικασία εξυγχρονισμού της συμφωνίας αυτής δεν βασίζεται σε οικονομικούς τόσο λόγους, όσο σε νομικούς, θεσμικούς και πολιτικούς περισσότερο λόγους, οι οποίοι δεν αποσαφηνίζονται και επακριβώς και αν έχετε ερωτήσεις ε, επ' αυτού θα προσπαθήσω να γίνω και λίγο πιο σαφής. Καθώς λοιπόν τα ζητήματα έχουν να κάνουν κυρίως με την νομική και την πολιτική προσέγγιση, θεωρώ ότι θα πρέπει να ασχοληθεί με το εξή ζήτημα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν θα πρέπει να συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ακολουθεί πιστά τα πρότυπα της Βορειοαμερικανικής Ζώνης Ελεύθερου Εμπορίου, της ναύτα, δηλαδή, στην εξωτερική οικονομική της ε, νομοθεσία και πολιτική, όπως έχει κάνει τα τελευταία χρόνια. Ξέρετε ότι ε, ο ευρωπαϊκός, η ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική τα τελευταία χρόνια έχει πειραστεί πάρα πολύ από την ναύτα. Οι εξωτερικές μας λοιπόν συμφωνίες ομοιάζουν όλο και περισσότερο με συμφωνίες τύπου ναύτα. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει να σε απασχολήσει το ζήτημα αυτό και να δείτε τελικά αν θα ήταν σκόπιμο να επιστρέψετε στις ε, παλιές, καλές, καλές ε, ευρωπαϊκές συμφωνίες σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρομαι τόσο στις ευρωπαϊκές όσο και στις ευρωμεσογειακές τέτοιες συμφωνίες. Οι παλιές καλές αυτές ευρωπαϊκές συμφωνίες ήταν δυναμικές πραγματικές συμφωνίες, ενώ συμφωνίες τύπου ναύτα είναι πραγματικά στάσιμες συμφωνίες. Η ρυθμιστική σύγκληση θα πρέπει να αποτελέσει επίση πραγματικό στόχο του εξυγχρονισμού τη συμφωνία αυτή. Δεν ξέρω αν το έχετε ιστοποιήσει αυτό το πράγμα. Οι παλαιότερε πατροπαράδοτε συμφωνίε Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν να κάνουν με ρυθμιστική σύγκληση. Φαίνεται να ξεκινάμε πάλι από την αρχή εδώ πέρα. Προκειμένου να πετύχουμε την κανονιστική αυτή σύγκληση, είναι πάρα πολύ σημαντικό οι εμπορικέ συμφωνίε να είναι δυναμικέ και να δημιουργούν το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θα μπορούσε πραγματικά να οδηγήσει σε αυτή την κανονιστική ρυθμιστική σύγκληση. Και δυστυχώ συμφωνίε τύπου ναύτα δεν οδηγούν σε κάτι τέτοιο. Ποιο είναι λοιπόν το πρότυπο το οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε για την νέα αυτή συμφωνία. Εσεί θα το αποφασίσετε αυτό. Ή η πατροπαρά του Ευρωπαϊκέ Συμφωνίε ή το μοντέλο το οποίο επιβάλλει αυτή τη στιγμή η Αμερική ή το μοντέλο το οποίο έχουμε ακολουθήσει τα τελευταία χρόνια στις διμερείς μας επενδυτικές και εμπορικές συμφωνίες. Για παράδειγμα, σε συμφωνίες που έχει συνάψει η Αμερική, οι Ηνωμένε Πολιτείε, δεν υπάρχει κανένα κεφάλαιο για την κυκλοφορία των εργαζομένων ενώ στο κοινοτικό δίκαιο έχουμε συγκεκριμένο τέτοιο κεφάλαιο και στο νοσιακό δίκαιο υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες, πολύ σημαντικοί κανόνες, οι οποίοι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο διεθνών διαπραγματεύσεων. Και αναφέρομαι πάντα στη μεταχείριση των αλλοδαπών εργαζομένων, οι οποίοι νομίμως εργάζονται στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για ποιο λόγο να μην έχουμε τέτοιες διατάξεις στη νέα αυτή συμφωνία. Αν εσείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματικά ανησυχείτε και από ό,τι φαίνεται ανησυχείτε για τα κοινωνικά ζητήματα και για την κοινωνική διάσταση των εμπορικών αυτών συμφωνιών, τότε ας μην γελιόμαστε. Μπορούμε να προσδώσουμε μια πραγματική κοινωνική υφή συμφωνία αυτή, προσδίδοντάς της ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για την μεταχείριση και την κυκλοφορία των λαδακών εργαζομένων. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει είναι αν θέλουμε να καλύψουμε ένα μείγμα πολιτικών. Εγώ ως εμπειρογνώμων στο ζήτημα αυτό είχα ασχοληθεί με το ζήτημα του μείγματο πολλών διαφορετικών πολιτικών, το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει και στη συμφωνία αυτή με το Μεξικό. Και αυτή η συμφωνία και οποιαδήποτε νέα συμφωνία θα καλύπτει τα περισσότερα ζητήματα τα οποία αποτελούν αυτή τη στιγμή αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ζήτημα όμως, πολιτικής, το οποίο τίθεται αυτή τη στιγμή είναι αν η νέα αυτή συμφωνία θα πρέπει να περιορίζεται μόνο σε αυτού του τομεί αποκλειστική αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τίθεται λοιπόν το ακόλουθο ερώτημα. Αν εσεί πραγματικά επιθυμείτε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να δραματίζει έναν παγκόσμιο ρόλο ισοδύναμο με αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας και περιορίζομαι στις δύο αυτές χώρες, τότε μπορεί από μόνη της η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο μέσω των αποκλειστικών της αρμοδιοτήτων όσον αφορά την εξωτερική πολιτική και το εμπόριο να κάνει κάτι τέτοιο πραγματικά αμφιβάλλω. Και αυτό διότι οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν κινούνται στο παγκόσμιο προσκήνιο με τέτοια δυναμικότητα έχοντας μόνο κάποιες ε, αρμοδιότητες. Οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Κίνα χρησιμοποιούν το ευρύτερο δυνατό σύνολο των αρμοδιοτήτων τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταφέρει να πείσει τα κράτη-μέλη να κάνουν κάποιες παραχωρήσεις όσον αφορά και τη δική τους αρμοδιότητα. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο, αν αναμίξουμε δηλαδή πολιτικέ που έχουν να κάνουν με αποκλειστική αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών, θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μια αποτελεσματική συμφωνία και θα καταφέρουμε να δώσουμε και μεγαλύτερη δυναμική στο ρόλο που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο παγκόσμιο προσκήνιο. Είναι πολύ σημαντικό τόσο για το Μεξικό όσο και για τα κράτη-μέλη να καταφέρουμε να κάνουμε μια αναφορά στην ανώτατη εκπαίδευση. Ξέρετε ότι το Μεξικό είναι μία από τις ε, χώρες στον κόσμο αυτό που έχει ένα από τα πιο φιλόδοξα προγράμματα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και ανώτης εκπαίδευσης και ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα υποτροφιών. Για ποιο λόγο λοιπόν στη νέα αυτή συμφωνία να μην εντάξουμε και ένα κεφάλαιο για την ανώτατη εκπαίδευση και κατά αυτόν τον τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει ένας ελκυστικός χώρος, μια ελκυστική περιφέρεια για τους ε, φοιτητές απανταχού στον πλανήτη. Είναι σίγουρο ότι αν ε, βάλουμε τέτοιο κεφάλαιο σε αυτή τη νέα συμφωνία, αυτό θα είναι και για το Μεξικό, αλλά και για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα ευρωπαϊκό κράτος το οποίο να μπορούσε να ανταγωνιστεί τις Ηνωμένε Πολιτείε, προς τις οποίες πηγαίνουν βέβαια οι περισσότεροι Μεξικανοί φοιτητέ. Πρέπει επίσης να δούμε ποιο είναι και το νέο καθεστώς όσον αφορά τις ξένες επενδύσεις. Έχουμε τη συμφωνία με τον Καναδά. Στη συμφωνία αυτή εξαιρείται η πολιτική αεροπορία και ο οπτικοακουστικός, οπτικοακουστικός με το τομέας. Και αυτό είναι λογικό, γιατί δεν επιτρέπεται εθνική μεταχείριση για τους δύο αυτούς τομείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις ευρωπαϊκές εκείνες εταιρείες που είναι κατεστημένες σε τρίτες χώρες. Αυτή τη στιγμή όμως στα πλαίσια των διμερών εθνικών συμφωνιών δεν αποκλείονται οι δύο αυτοί τομείς. Τι θα γίνει λοιπόν με τους δύο αυτούς τομείς, οι οποίοι καλύπτονται όπως σας είπα από διμερείς επενδυτικές συμφωνίες των κρατών μελών οι οποίοι όμως δεν συνάδουν αυτή τη στιγμή με τους κοινοτικούς κανόνες που υφίστανται για τις ξένες επενδύσεις. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να ασχοληθούμε με το ζήτημα αυτό που είναι πολύ πιο ουσιαστικό από τα ζητήματα της διαιτησίας ή των αρμόδιων δικαστηρίων. Το Μεξικό δεν θα πρέπει να στερείται στα πλαίσια μιας Ευρωπαϊκής Συμφωνίας δικαιώματα τα οποία έχει στα πλαίσια διμερών συμφωνιών που έχει συνάψει με, μονομένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κάτι ακόμα. Ένας κίνδυνος, ένας πολιτικός κίνδυνος να υιοθετήσει τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση μία αμυντική στάση στα πλαίσια της αναθεώρησης αυτής της συμφωνίας. Γιατί να γίνει κάτι τέτοιο θα μου πείτε, μα διότι το Μεξικό έχει ήδη ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις για μια πολύ φιλόδοξη εμπορική και επενδυτική συμφωνία που είναι το Trans-Pacific Partnership, η εταιρική σχέση για τον ειρηνικό. Προτίθεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να αποδειχθούν το βαθμό φιλοδοξίας που υπάρχει σε αυτή την εταιρική σχέση για τον ειρηνικό. Αν διαβάζετε το κείμενο της συμφωνίας αυτής, το κείμενο είναι ήδη, έχει ήδη δημοσιευτεί, τότε πραγματικά θα συνειδητοποιήσετε ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια αυτή. Ας μην ξεχνάμε ότι το Μεξικό θα ξεκινήσει από αυτό το σημείο φιλοδοξίας για το Μεξικό, αυτή η εταιρική σχέση για τον ειρηνικό θα αποτελέσει το σημείο αναφορά. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ εύκολα θα βρεθεί σε μια αμυντική στάση και όχι σε μια επιθετική στάση όπω θα έπρεπε. Γι' αυτό διότι θα φανεί πάρα πολύ γρήγορα ότι το Μεξικό είναι πολύ πιο φιλόδοξο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το περιεχόμενο, το πεδίο εφαρμογή και του στόχου αυτή τη συμφωνία. Αυτά είχα να Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω πως θέσετε κάποια δύσκολα ερωτήματα. Τώρα θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Ε, David Martin. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον εμπειρογνώμονα για αυτήν την ενδιαφέρουσα παρουσίαση και τους δύο εμπειρογνώμονες να ευχαριστήσω για πολύ ποιοτική δουλειά. Ε, ως ε, σκιώδης, εκπρόσωπος του σκιώδου συζητητού θα διαβάσω μία δήλωσή του. Δυστυχώς ε, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να έρθει γιατί συζητά για το θέμα των θεωρήσεων με εκπροσώπους του Καναδά. Είναι λοιπόν η κατάλληλη στιγμή διότι από τότε που άρχισαν οι διαπραγματεύσεις ο πρώτος κύκλος έγινε στις Βρυξέλλες νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα. Συζητήθηκαν διάφορες πτυχές πολιτικής κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων. Θα ήθελα όμως να πω το εξής. Ο εξυγχρονισμός του πυλώνα εμπορίου της συμφωνίας με το Μεξικό είναι αναγκαίο παρά ε, κάτι ε, απλά διευκολυντικό. Ο εμπορικός πυλώνας και, το, η νέα γενιά εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνδέονται άμεσα. Το βλέπουμε και από το κείμενο της Συμφωνίας ΣΥΤΑ, αλλά και άλλες ε, συμφωνίες, την TPP, τη Συμφωνία με την Κολομβία και το Περού κτλ. Αυτό δείχνει ότι χρειάζεται βελτίωση, όχι μόνο για την πρόσβαση στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών, όχι μόνο για την συνοχή, για την διευκόλυνση του εμπορίου, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις γεωγραφικές ενδείξεις και τις δημόσιες προμήθειες, αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει σχέση ανάμεσα στα ανθρώπινα δικαιώματα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και το εμπόριο. Αυτό μέχρι στιγμή δεν διαφαίνεται στι παγκόσμιε εμπορικέ συμφωνίε. Δεν υπάρχει ούτε ένα κεφάλαιο για την βιώσιμη ανάπτυξη. Και αυτή είναι μια ιδανική ευκαιρία να γίνει συμφωνία, μια σύγχρονη συμφωνία με ε, προηγμένες και αποτελεσματικές διατάξεις, για παράδειγμα για την ε, βιώσιμη ανάπτυξη και κατά της διαφθοράς έχει στρατηγική σημασία και, και τα δύο συμβαλόμενα μέρη να αναγνωρίσουν το πόσο σημαντική είναι μια τέτοια συμφωνία. Το Μεξικό είναι ο πιο σημαντικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Και ε, αυτά συνοπτικά είναι τα λόγια του σκιώδου συζητού και εγώ να ζητήσω συγγνώμη διότι πρέπει να γυρίσω πίσω στο ε, Ηνωμένο Βασίλειο για να προσπαθήσω να, ε, του, να κάνω εξτρατεία κατά του Brexit. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πάπλο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αναμφίβολα είναι ιδιαίτερα κατάλληλη η στιγμή για αυτή την έκθεση που μας παρουσιάστηκε. Γιατί οπωσδήποτε θα συμβάλλει ούτως ώστε αυτές οι διαπραγματεύσεις Ένωσης Μεξικού να είναι οι καλύτερες δυνατές. Είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να υπάρξει ενημέρωση του εμπορικού πυλώνα της εταιρική ε, σχέσης, της Συμφωνίας Σύνδεσης της Ένωσης Μεξικού, γιατί όταν ε, συνήφθη αυτή η συμφωνία ήταν πολύ διαφορετικές συνθήκες και οι συμφωνίες που διαπραγματεύεται τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτους ε, πολύ λίγη σχέση έχουν με αυτό που γινόταν τότε. Πρέπει λοιπόν να εξυγχρονιστεί και στη στηρίζω την προσπάθεια αναμφίβολα, χωρίς επιφυλάξεις. Αν καταλήξουμε σε μια σωστή, ισορροπημένη συμφωνία, θα ε, είναι αμοιβαία επωφελής. Είναι λοιπόν σκόπιμη αυτή η συζήτηση σίγουρα θα ωφελήσει ε, αμοιβαία τους ε, συμπολίτες μας και τους πολίτες του Μεξικού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ισκά Κέλλερ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Έχω κάποιες ερωτήσεις για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βασισμένη στην ε, μελέτη που μόλις είδαμε, αλλά και εσείς αν θέλετε να μου απαντήσετε. Για λοιπόν, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ είστε. Ακούσαμε την παρουσίαση και κοιτάζοντας τη μελέτη βλέπω ότι πολλοί στο Μεξικό δεν γνωρίζουν πολλά ή δεν είναι και ιδιαίτερα υπέρ και εκείνοι που είναι υπέρ δεν θέλουν να αλλάξουν πολλά. Αυτό λοιπόν πρέπει να μας κάνει να προβληματιστούμε. Ποιο είχε την αρχική ιδέα για να εξυγχρονιστεί η συμφωνία. Θεωρείτε πως είναι καλή ιδέα να προχωρήσουμε αν κανείς δεν το θέλει. Για μας, δεδομένου ότι έχουμε πάρα πολλές συμφωνίες και πάρα πολλή δουλειά, δεν ξέρω αν θα ωφελούσε να είχαμε ακόμα περισσότεροι, εφόσον κανείς δεν θέλει αυτή τη συμφωνία. Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν κατάλαβα καλά από αυτά που άκουσα, είναι να μειωθεί η φτώχεια και οι ανισότητες. Όμως, από τότε που υπεγράφει αυτή η Παγκόσμια Συμφωνία, βλέπουμε αύξηση και των δύο. Γι' αυτό λοιπόν δεν νομίζω πως μπορώ να είμαι πολύ αισιόδοξη για το ότι θα μειωθούν η φτώχεια και η ανισότητα. Και μία ερώτηση και προς τους συντάκτες τη μελέτη και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το όλο θέμα του οργανωμένου εγκλήματο. Είναι ένα σημαντικό πρόβλημα στο Μεξικό και συνδέεται και με ξέπλυμα χρήματο. Βλέπουμε ότι υπάρχει τέτοιο πρόβλημα και στις πορικέ σχέσει ανάμεσα στο Μεξικό και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι πολύ δύσκολο να ε, μην υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Και μάλιστα η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι πολύ διαδεδομένη και έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στο Μεξικό. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται με τις ε, συμφωνίες που ε, στηρίζουν έστω και με έμεσο τρόπο αυτές τις παράνομες δραστηριότητες και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη ροή παράνομου χρήματος προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, για το κοινό συμβούλιο που προβλέπεται σύμφωνα με την ε, συμφωνία με το Μεξικό. Υπάρχει κάποιο σχέδιο να ε, υποβάλλεται εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις εργασίες του. Διότι δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Και κάτι πάνω στη μελέτη. Αναφέρθηκε αρκετές φορές ότι καλό θα ήταν να υπάρχει ένα υποχρεωτικό ένας υποχρεωτικός χαρακτήρας για μέτρα που δεν είναι αμυγός οικονομικά. Ποιες θα λέγατε πώς είναι οι προτεραιότητες έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα ε, τέτοιο σύστημα για τις οικονομικές δραστηριότητες. Τι θα προτείνατε, τι θεωρείτε πως ε, έχει προτεραιότητα. Ευχαριστώ. Ο Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να υποβάλω κάποιες ερωτήσεις και για τη μελέτη, αλλά και για τη διαδικασία που θα ακολουθήσουμε για αυτόν τον πυλώνα ελεύθερου εμπορίου, στα πλαίσια μάλλον αυτή της παγκόσμια συμφωνία. Νομίζω καταρχάς Πώ είναι θετικό ότι οι συντάκτες της μελέτης αναγνώρισαν ε, το ρόλο μας και σε αυτό το παγκόσμιο πλαίσιο. Το πώς θα μπορούσαν να αναπτυχθούν οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μεξικού και πώς θα μπορούσε να εξυγχρονιστεί η συμφωνία. Θα ήθελα όμως περισσότερες λεπτομέρειες, πιο συγκεκριμένα. Ναύτα, TPP, αυτές οι συμφωνίες, οι ε, δεσμευτικές ε, διατάξεις, αλλά κοιτάζοντας και τις γενικότερες πτυχές ε, που διέπουν διεθνείς συνεργασίες σε όλες τις συμφωνίες και με άλλες χώρες. Αυτό που δεν είδα είναι μια πιο εις βάθος ανάλυση σχετικά με τις προϋποθέσεις για αυτόν τον εξυγχρονισμό του εμπορικού πυλώνα μέσα στο Μεξικό. Μας είπατε ότι υπάρχουν ακόμα πολλά ερωτηματικά, ότι δεν είναι σίγουρο αν το επιθυμούν. Μας μιλήσατε για διαφορές δημοσκοπήσεις, όμως τι συμβαίνει ακριβώς μπορεί η οικονομία του Μεξικού να εξελιχθεί και εκείνη στις ε, σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να φτάσει σε τέτοιο σημείο ώστε να είναι δυνατή η υπογραφή μιας τέτοια εμπορική συμφωνίας. Υπάρχουν πολλά προβλήματα στις ε, εξελίξεις εντός του Μεξικού όπως ε, ανέφερε και η συνάδελφος, φτώχεια, ανισότητα, έγκλημα, το έγκλημα αυξάνεται. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η κοινωνία είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό για τους οικονομικούς εταίρους του Μεξικού. Και μπορούμε να διαχωρίσουμε τις εμπορικές επιχειρήσεις από αυτές τις εξελίξεις ε, στη χώρα. Έπειτα, το ξέπλυμα χρήματος αναφέρθηκε και από την Σκά Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω όμως εάν αναφέρεστε στην χρηματοοικονομική διάσταση αυτού και τι σημαίνει αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα από χρηματοοικονομικής πλευράς. Η νομοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητε είναι ένα μόνο μέρος του προβλήματος. Ο Ντέιβιτ Μάρτιν ανέφερε και την βιώσιμη ανάπτυξη. Πώς λοιπόν θα συμφωνήσουμε με τους εταίρους μας στο Μεξικό για τα διάφορα ε, κοινωνικά, οικολογικά κριτήρια σε αυτό το κεφάλαιο, τα οποία φυσικά και πρέπει να αναφερθούν, να συμπεριληφθούν και να προβλέπονται δεσμευτικές διατάξεις. Δεν νομίζω ότι το Μεξικό είναι έτοιμο για δεσμευτική συμφωνία. Ακόμα και εμείς στην Ευρώπη συζητούμε εάν θα πρέπει να έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, να υπάρχουν μηχανισμοί επιβολής ε, της συμφωνίας. Υπάρχει και η γνωμοδότηση της Επιτροπής μας για τη στρατηγική εμπόριο για όλους και επίσης η παρακολούθηση των περιβαλλοντικών κοινωνικών πτυχών της πολιτικής. Και φυσικά έχει λάβει θέση η Επιτροπή μας, είναι θετικά προσκύμενη. Αναφέρθηκαν και οι ε, Παγκόσμιες Συμφωνίες Ελεύθερου Εμπορίου αλλά νομίζω πως ενδεχομένως είναι θέμα εντολής. Νομίζω οι διαπραγματεύσεις προβλέπονται για το φθινόπωρο φέτος. Αναρωτιέμαι λοιπόν τι χρονοδιάγραμμα θα έχουμε εμείς. Διότι το Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει τη δική του θέση προτού δοθεί εντολή. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να διαμορφώσουμε θέση πριν την εντολή, η οποία εντολή πρέπει να είναι δημόσια ευθύ εξ αρχή. και πρέπει να ζητήσουμε η διαδικασία να είναι διαφανής. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να υπάρχει μια ε, ανταλλαγή απόψεων με όλους τους φορείς για όλα τα ε, ε, θέματα, αλλά πρέπει να μας αφήσετε αρκετό χρόνο για να κάνουμε τη δουλειά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Τι έχει να πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για όλες αυτές τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να σας απαντήσω και να σας πω πώς έχουν τα πράγματα όσον αφορά την ακολουθητέα διαδικασία. Πρώτον, ξεκινάμε τις διαπραγματεύσεις αυτές με στόχο να είμαστε ως το δυνατόν πιο διαφανείς και θέλουμε να είμαστε απόλυτα διαφανείς βέβαια και απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και συμφωνούμε απόλυτα μαζί σας ότι όντως θα ήταν σκόπιμο η διαπραγματευτική εντολή που θα λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το Συμβούλιο να είναι δημόσια, αλλά αυτό βέβαια είναι απόφαση Συμβουλίου, όπως ξέρετε. Συμφωνούμε πάντως από αυτού απόλυτα μαζί σας. Τώρα, αναφερθήκατε σε μία εμπορική συμφωνία και όντως υπάρχει εμπορική συνιστόσα σε αυτή τη συμφωνία. Αλλά μην ξεχνάμε ότι με το Μεξικό έχουμε μία συνολική συμφωνία. Εμείς δεν εξυγχρονίζουμε απλώς μία εμπορική συμφωνία, αλλά το σύνολο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης που έχουμε με το Μεξικό. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι στα πλαίσια της επικαιροποίησης αυτής θα ασχοληθούμε και με τα εμπορικά ζητήματα είναι και αυτά μέρος του όλου πακέτου αν θέλετε, αλλά θα ασχοληθούμε και με όλες τις άλλες πολιτικές σχέσεις που έχουμε το Μεξικό και με όλες τις άλλες μορφές συνεργασίας. Και σίγουρα θα καλύψουμε και τη δυνατότητα να κινηθούμε σε άλλους τομείς όπως η ανώτατη εκπαίδευση που ανέφερε ο Ραμόν Τορέντε πριν από λίγο. και θα κινηθούμε σε αυτό το δρόμο, ιδίως όσον αφορά το κεφάλαιο εκείνο που έχει να κάνει με την ε, πολιτική συνεργασία. Για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή θέλουμε να κάνουμε τον εξυγχρονισμό αυτό. Το, το ρώτησε αυτό η Σκά Κέλλερ. Κοιτάξτε, είναι πολιτική απόφαση που έχει ληφθεί σε υψηλότατο επίπεδο. Υπάρχει λοιπόν η απαραίτητη πολιτική βούληση ανάμεσα στους ε, αρμόδιους ηγέτες το 2013 λήφθη η πρώτη αυτή απόφαση και επικαιροποιήθηκε πέρυσι στην τελευταία σύνοδο που είχαμε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μεξικού, όπου και οι δύο πλευρές είπαν ότι προτίθενται να προχωρήσουν με τον εξεχρονισμό αυτή τη συμφωνία. Ουσιαστικά εμεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρινόμαστε σε ένα πολιτικό αίτημα το οποίο έχει έρθει από το υψηλότατο δυνατό επίπεδο. Και επίση, ανταποκρινόμαστε και στι απαιτήσει τη κοινωνία των πολιτών. Όταν ξεκινούσαμε τις διαπραγματεύσεις αυτές, γενικά όταν κάνουμε εμπορικές διαπραγματεύσεις, κάνουμε παράλληλα και μια δημόσια διαβούλευση. Επί της συμφωνίας αυτής είχαμε πολύ θετική ανταπόκριση και από τις επιχειρήσεις, αλλά και από την κοινωνία των πολιτών και από μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Όλοι αυτοί συνέβαλαν με τρόπο ιδιαίτερα επικοδομητικό για μας και καταφέρουμε κατά αυτόν τον τρόπο να κάνουμε μια σωστή αξιολόγηση των διαπραγματεύσεων που θα πρέπει να κάνουμε και ποιες ήταν οι επιπτώσει αυτών των διαπραγματεύσεων. Και έτσι φτάσαμε στο επόμενο βήμα της ε, αξιολόγησης αυτής, η ε, αξιολόγηση αντικτύπου, βιώσιμου αντικτύπου, την οποία αξιολόγηση θα μπορέσετε και εσείς βέβαια να συμμετάσχετε και θα γίνει στις αρχές, ελπίζω, του επόμενου έτους. Και θα εξετάσουμε και τα υπόλοιπα ζητήματα που δικαίω θέσατε, ποιε ήταν οι επιπτώσει όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, ποιε είναι οι επιπτώσει στα εργασιακά δικαιώματα, ποιο είναι ο αντίκτυπο στο περιβάλλον και το καθεξής. Στη συνέχεια, σε σχέση με την ομοιοποίηση παράνομων ε, εσόδων, ακούσαμε διάφορες ερωτήσεις επ' αυτού συμφωνούμε και συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες σας. Είναι σημαντικό οι εμπορικές συμφωνίες να συμβάλλουν στη χρηστή διακυβέρνηση και μέσω αυτό να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ζητήματα όπως η διαφθορά. Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι έχουμε μια εμπορική πολιτική που θα διέπεται από συγκεκριμένε αρχές. Βλέπετε όμως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι όντως η εμπορική πολιτική θα πρέπει να συμβάλλει για όλα αυτά τα ζητήματα. Αυτό το βλέπετε και στην ακοίνωσή μας εμπόριο για όλους. Και είπαμε ότι θέλουμε να προωθήσουμε τα διεθνή πρότυπα της διαφάνειας και της χρηστής διακυβέρνησης στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας. Πώς θα γίνει όμως τώρα κάτι τέτοιο στην πράξη και πώς μπορεί αυτό να συνδυαστεί με το ότι αυτή τη στιγμή θέλουμε να έχουμε την, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στους α, επιμέρους τομείς συμφωνίας και πώς μπορεί η πρόθεσή μας αυτή να συνδυαστεί με το ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς ή του ξεπλήματος ε, βρώμικου χρήματος αντιμετωπίζεται ήδη από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών ή αντιμετωπίζεται από υπηρεσίες του ΟΣΑ και εμείς δεν θέλουμε σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργήσουμε εδώ πέρα μία επικάλυψη. Είναι πάντως σημαντικό οι συμφωνίες μας αυτές να μην λειτουργούν μεμονωμένα, αποκομμένα, αλλά να μπορούν να συμπληρώνουν τις διαδικασίες αυτές που έχουν ξεκινήσει τα Ενωμένα Έθνη και ο ΩΣΑ. Θα είμαι σύντομο, Πρόεδρε. Έγινε μια πρώτη συζήτηση με το Μεξικό την Δευτέρα και την Τρίτη. Δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Είμαστε, αν θέλετε, σε ένα πρώτο στάδιο, κοντά στην αρχή, αλλά έχουμε προχωρήσει και για πρώτη φορά καταφέραμε να δούμε ποια είναι η εμπειρία που έχει η μεξικανική πλευρά από το GPP όσον αφορά την καταπολέμηση της ε, διαφθοράς. Και ολοκληρώνω στο σημείο αυτό, όντως δεν έγινε καμία αναφορά όσον αφορά τις αποφάσεις του Κοινού Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεξικού. Όντως ε, δεν συνεδρίασε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα το Κοινό αυτό Συμβούλιο, ακριβώ επειδή θέλαμε να δούμε πώς θα καταφέρουμε να επικαιροποιήσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη συμφωνία. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα το λόγο πάλι έχει ο συντάκτης μελέτης για 5 λεπτά. Εάν ήμουν εδώ ως εκπρόσωπος της Κομισιόν, δεν θα μπορούσα να απαντήσω καλύτερα από ότι απάντησε ο κύριος Τζόρκιτς. Συμφωνώ λοιπόν με πολλά από όσα είπε, γιατί ήταν πολύ ειλικρινής έναντί σας. Υπήρξε μια πολιτική απόφαση, τονίζω, πολιτική απόφαση. Αυτό είναι σαφές. Εφόσον λοιπόν έχει ληφθεί η πολιτική απόφαση να υπάρξει εξυγχρονισμός της συμφωνίας, ενημέρωση της συμφωνίας, οι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, θα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. από τη διαπραγματευσή. Ο κύριος Γιόρκετς μας είπε ότι η νέα συμφωνία, η οποία θα είναι ευρεία, θα υιοθετηθεί κατά πολύ προσέγγιση της βέλτιστης ε, προσπάθειας, του βέλτιστου εγχειρήματος. Λοιπόν, με βάση την ε, μελέτη μας, δεν είναι το Μεξικό που ε, ενδιαφέρεται τόσο πολύ. Το Μεξικό θα μπορούσε να έρθει εδώ, να αναφερθεί στην, ε, στο TPP και θα μπορούσαν ε, να έχουν ένα παρόμοιο, μια παρόμοια συμφωνία διατλαντική. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορούσε να την υπογράψει. Άρα τα προβλήματα δεν τα έχει το Μεξικό για αυτή τη διαπραγμάτευση, αλλά εμείς. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Δεύτερο θέμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί θέματα που μπορούν να λυθούν ε, ενδοενωσιακά πρέπει να εξαχθούν μέσω των διαπραγματεύσεων με το Μεξικό. Αν θέλετε να προστατεύσετε τόσο πολύ τα συμφέροντα της ανθρωπότητας, εάν θέλετε νέα νομοθεσία για το οργανωμένο έγκλημα και το ξέπλυμα χρήματος, δεν χρειάζεται συμφωνία με το Μεξικό για να αλλάξετε την νομοθεσία. Το πρόβλημα είναι ότι κατά τη λογική της μελέτης μας κανείς δεν θέλει. Κανείς στην Ευρώπη δεν θέλει να αλλάξει αυτή η νομοθεσία. Και αν δεν θέλει κανείς, πώς θα απαιτήσετε να αλλάξει το Μεξικό την νομοθεσία του. Τελειώνω, τελειώνω. Άλλο ένα σημείο. Ο Κάρλος Λίμ είναι ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου. Ελέγχει μία από τη μεγαλύτερη εταιρεία ε, υπηρεσιών στην Ισπανία, την FCC. Και με βάση τη διμερή συμφωνία για τις επενδύσεις μεταξύ Ισπανίας και Μεξικού, η FCC, την οποία ελέγχει ο Κάρλος Σλιμ, θα μπορούσε να αγοράσει την αεροπορική εταιρεία Βούλινγκ της Ισπανίας. Αλλά σύμφωνα με τον κανονισμό για τις αεροπορικές άδειες δεν μπορεί την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Γιατί αν το FCC αγοράσει την Vueling, η Vueling θα, έχασε, θα έχανε την άδειά της. Γιατί θα ήταν υπό μεξικανικό έλεγχο. Αυτός είναι ένας κανονισμός που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και ισχύει. Γιατί λοιπόν το Μεξικό, γιατί να παραιτηθεί ενό δικαιώματό του μέσω των διαπραγματεύσεων, δεν το έχει βεβαίω επικαλεστεί μέχρι τώρα. Αλλά μέσω τη διμερού συμφωνία που έχει το Μεξικό με την Ισπανία, έχει αυτό το δικαίωμα. Τέτοιου τύπου θέματα είναι ουσιώδη για το τι θα σημάνει ο εξυγχρονισμό, για το τι σημαίνει ότι θέλουμε μια φιλόδοξη στρατηγική σχέση. Αυτά είναι ουσιώδη θέματα που θα συζητηθούν στη διαπραγμάτευση και οι φίλοι μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν πολλή δουλειά μπροστά τους και θα έχουν μεγάλες δυσχέρειες για να απαντήσουν εάν το Μεξικό θέσει αυτά τα θέματα. Αυτά πρέπει να σας απασχολήσουν. Αυτά και ορισμένα άλλα τα οποία τα τονίζουμε στην έκθεσή μας και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω θα συνεχίσουμε τον προβληματισμό μας πριν τη συμφωνία και θεωρώ ότι η μελέτη σας θα επηρεάσει πολύ θετικά ε, τις εργασίες μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον πρεσβευτή του Μεξικού που ήρθε. Σημείο 19 της ημερήσιας διάταξης είναι τα διάφορα. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι στις 21 Ιουνίου θα έχουμε μία συζήτηση για τις διαφορές ανάμεσα στις ε, συμφωνίες εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΕΖΕΣ. Μετά την ψηφοφορία στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 23 Ιουνίου θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Μπορεί να έχουμε να συζητήσουμε και εμπορικές συμφωνίες με το Ηνωμένο Βασίλειο. Επόμενη συνεδρίαση, μάλλον η συνεδρίαση αυτή θα γίνει στο α3G2. Επόμενη συνεδρίαση στις 30 Ιουνίου. Αυτά, καλό Σαββατοκύριακο.